Sit down, please. Καθίστε παρακαλώ. Buongiorno a tutti. La Καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Σήμερα το πρωί θα γίνει η εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των διατάξεων του κανονισμού μας και όχι βάσει αποφάσεων και εξωτερικών προτάσεων. Πρόκειται για ελεύθερο κοινοβούλιο και αυτόνομο κοινοβούλιο. Να σας ανακοινώσω ότι έλαβα βάση ε, των διατάξεων του κανονισμού τις ακόλουθες υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Σκά Κέλλερ. Ο κύριος Σύρα Ρέγκο. Ο κύριος Ντάβιτ Μαρία Σασόλη. Και ο κύριος Γιάνν Ζαχαντή. Όλοι οι υποψήφοι επιβεβαίωσαν ότι αποδέχονται την υποψηφιότητά τους και πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία θα δώσω εν συντομία το λόγο σε κάθε έναν από τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Ο καθένας θα έχει στη διάθεσή του 5 λεπτά για να κάνει την παρέμβασή του. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σκακέλερ. Dear of the European Parliament. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι και βασικότερο αγαπητοί Ευρωπαίοι πολίτες. Πριν από πέντε εβδομάδες οι Ευρωπαίοι πολιτές άσκησαν το δικαίωμά τους και μας εξέλεξαν ως αντιπροσώπους τους. Ασκήσατε το δικαίωμά σας για να διαμορφώσετε το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που εμπιστευτήκατε αυτό το θεσμικό όργανο. Θα μας δώσατε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι ζωντανό. Εσείς, οι ψηφοφόροι, απαντήσατε τη, στην ε, διχαστική ρητορική της λαϊκιστικής δεξιάς με το ξεκάθαρο μήνυμά σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι εκλογές αυτές είδαν αυξημένη προσέλευση των ψηφοφόρων, κάτι το πολύ ενθαρρυντικό, αλλά αυτό σημαίνει και αυξημένη ευθύνη για εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρη στους ψηφοφόρους έχουμε μια ισχυρή εντολή για να αποφασίσουμε τώρα για το μέλλον της Ευρώπης και για να λογοδοτούν σε εμάς τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν. Και έχουμε λάβει εντολή να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο. Και εγώ λέω ας ενισχύσουμε το Κοινοβούλιο σήμερα και ας γίνει αυτό με το να εκλέξουμε μία πρόεδρο η οποία θα ενσαρκώνει την ανεξαρτησία του θεσμικού μας Ιδρύματος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε η Προεδρία του Κοινοβουλίου να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε παλαιού τύπου παζάρια στο Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Εν ώψη της κλιματικής κρίσης, κοινωνική ανισότητας και των διεθνών αντιπαραθέσεων. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ. Αλλά πάντα εμείς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν ήμασταν επιτυχεί στο να ερχόμαστε σε επαφή με τους πολίτες και να τους πείσουμε ότι αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που τους απασχολούν. Ω πρόεδρο, θα ήθελα να ανανεώσω αυτή την εμπιστοσύνη και να διασφαλίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ο χώρο όπου οι πολίτε συζητούν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συζητήσει για το μέλλον τη Ευρώπη με αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, με πρόεδρου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε. Γιατί να μην αλλάξουμε κατεύθυνση και να λέμε να ανοίξουμε το Κοινοβούλιο, να συζητήσουμε το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση με του πολίτε, με την κοινωνία των πολιτών, με του ανθρώπου που διαμορφώνουν την ήπειρό μα σήμερα. στο Κοινοβούλιο σαφώς υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, το κράτο δικαίου. Και ω πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα ήθελα να είμαι η πρέσβυρα για αυτές ακριβώς τις αξίες και αρχέ. Και για να είμαστε αξιόπιστοι και ως θεσμικό όργανο θα πρέπει κάθε μέρα να εργαζόμαστε για να ακολουθούμε αυτέ τι αρχέ που ζητάμε και από άλλου να ακολουθήσουν. Είτε μιλάμε για διαφάνεια, είτε για ισότητα των φίλων συμπερίληψη, δικαιώματα των εργαζομένων και μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος. Και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο ιστορικό επίδευμα της Υπήρου μας. Έχει διασφαλίσει ειρήνη, φιλία και ευημερία στην, σε μια Ήπειρο η οποία είχε πολέμους και μίσος ως ερετοί ευρωβουλευτές. Έχουμε μια κοινή ευθύνη να τιμήσουμε και να υπερασπίσουμε αυτό το ιστορικό επίτευγμα που κληρονομήσαμε. Και εγώ γεννήθηκα σε μια χώρα η οποία ήταν διχασμένη από το σιδηρούν παραπέτασμα. Ήμουν στα σύνορα Πολωνίας και Γερμανίας και έχω δει με τα μάτια μου το τι σημαίνει να ενώνει η Ευρώπη τους ανθρώπους, να ξεπερνά τα σύνορα και στα μυαλά και στο έδαφος. Και έχω δει επίσης και την προσωπική ευθύνη να υπερασπιστούμε αυτήν την ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε και το θάρρο να την αλλάξουμε προ το καλύτερο. Και ω το μοναδικό θεσμικό όργανο το οποίο είναι απευθεία αιρετό από του πολίτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν ρόλο κλειδί σε αυτό το άλμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια παλεύει για να υπερασπιστεί και να αυξήσει τα δικαιώματά του, γιατί αυτό σημαίνει να αυξήσει τα δικαιώματα και την εκπροσώπηση των πολιτών, των πολιτών που μας ψηφίζουν και μας στέλνουν εδώ πέρα. Και για να συνεχιστεί αυτή η δουλειά είμαι σήμερα υποψήφια και ελπίζω να μου κάνετε την τιμή να με εκλέξετε πρόεδρο του κοινοβουλίου αυτού. Και θα σας είμαι ευγνώμων. la parola. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σιραρέγο. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ μια ομάδα η οποία υπερασπίζεται τα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και ιδίως των εργαζομένων. Παρουσιάζουμε αυτή την υποψηφιότητα από την αρχή, ενώ κάποιες ομάδες και κυβερνήσεις της Ευρώπης παζαρεύουν ε, τις καρέκλες, η ζωή και το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων ε, εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε σε αυτό το κοινοβούλιο. Γι' αυτό για μα είναι απαραίτητο να μιλήσουμε σε ποια πλευρά πλευρά θα είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα επόμενα έτη θα συνεχίζει να είναι πλάι στα λόμπι και στις πολυεθνικές. Θα είναι από την πλευρά της Ευρώπης των τυχών και θα συνεχίσει να τροφοδοτεί το τέρας του νεοφασισμού. Ή όπω θέλουμε εμείς ε, θα είναι στην πλευρά των λαών, των εργαζομένων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς, οι γυναίκες, περασπίζουμε ένα κοινοβούλιο που απαντά στις ανάγκες των λαών μας, ε, που βασίζεται στη λαϊκή Κυριαρχία και που εργάζεται για να σταματήσει να βασίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζομένων η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι οικονομικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλαν σε δύσκολη θέση ολόκληρε χώρε, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα το ε, είδαμε αυτό, υποφέραμε, προκαλεί δεινά ανεργία, επισφάλεια και ανισότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πολιτικές μας στέλνουν σε μια ζωή χωρίς ελπίδα και χωρίς μέλλον. Και όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο. Αυτές οι πολιτικές και το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο ευθύνονται επίση για την κοινωνική και ε, κλιματική κρίση του πλανήτη. Το να αρνούμαστε είναι ε, να έχουμε ψευδεστήσεις. Ε, αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται δεν θα λύσει ένα πρόβλημα που αρχίσαμε να βιώνουμε σε κάθε κράτος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτό να είναι ένα από τα κυρία θέματα που θα προσεγγίσει το Κοινοβούλιο και γι' αυτό σας ζητάμε να υποστηρίξετε την πρότασή μας για να δημιουργήσουμε μια ειδική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή. Είναι απαραίτητο τώρα. Όμως ε, Ακόμη περισσότερο, οι νοφιλελεύθερες πολιτικές είναι αυτές ε, που τροφοδοτούν το τέρας του φασισμού. Εδώ ε, βρίσκεται η ακροδεξιά και ε, εδώ υιοθετεί κάποιες ρατσιστικές, αντισεξιστικές πολιτικές. Δεν θέλουμε το Κοινοβούλιο να αιτιολογήσει αυτή τη ρητορική μίσωση ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν κάποιες ε, μέρες ε, ε, συνελήφθη Καρόλα Ρακέτε, μια ηρωίδα που σώζει ζωές στη Μεσόγειο παρά το ότι ο Σελβίνη θέλει να ποινικοποιήσει το έργο της. Προτείνουμε αυτό το κοινοβούλιο να δώσει νομική κάλυψη σε κάθε άνθρωπο που διώκεται επειδή σώζει ζωές. Και εγώ που προέρχομαι από το Νότο, από την χώρα που απεργεί την ημέρα των γυναικών. Εμείς ξέρουμε ότι ο φεμινισμός ε, είναι μια δύναμη που θα σταματήσει το φασισμό Ξέρουμε ότι όλα θα τα ανατρέψει και θα προτείνει μια νέα κοινωνία. Προτείνουμε στι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσουν να ε, μα εξαπατούν. Εμεί οι γυναίκε θέλουμε φεμινιστικέ πολιτικέ, όχι ποσοστώσει. Θέλουμε ε, να συμμετέχουμε στην πολιτική και θα απαιτήσουμε φεμινισμό να είναι παρόν στο in agenda των θεσμικών οργάνων, όχι σαν ετικέτα, αλλά σαν ένα καλούπι πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τι κοινωνίε μα. Ε, θέλουμε να καταστεί ορατή η ιστορία των αόρατων γυναικών. Ε, πάνω στους ώμους τους οικοδομήθηκαν οι χώρες μας. Εμείς οι γυναίκες είμαστε που θέτουμε τα θεμέλια της κοινωνίας μας εδώ ε, ξέρουμε ποιο πλευρό λαμβάνουμε, υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών, των εργαζομένων, που κερδίζουν το ψωμί τους με την προσπάθειά τους. Γι' αυτό θέλουμε μια αδελφική και αντιφασιστική Ευρώπη. Ε, ξεκίνησε από Ισπανούς Ρεπουμπλικάνους η γαλλική αντίσταση. Είχαμε και τον Μανώλη Γλέζο, ο οποίος έβγαλε τη σημαία των Γερμανών από την Ακρόπολη στην Αθήνα ε, και επίσης ξεκίνησε από τους Ιταλούς Παρτιζάνου του Μπελατσάου που αντιστάθηκαν στο Μουσολίνι. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε, όμως διεκδικούμε και τους σημερινούς αγώνες και αναγνωριζόμαστε σε αυτούς. Η αξιοπρέπεια ε, των ακτιβιστών από την Open Arms και το Sea που σώζουν άτομα κατά του φρουρίου Ευρώπη. Αναγνωρίζουμε τις κινητοποιήσεις των νέων που υπερασπίζουν ε, το δικαίωμα τους ε, να ζουν σε αυτό αυτό πλανήτη, η Ευρώπη με το φεμινισμό θα αλλάξει τα πάντα. Γι' αυτό δεν μεσμόμαστε. Αυτό το κοινοβούλιο οικοδομήσει μια ειρηνική, αλληλέγγυη Ευρώπη και δεν θα αφήσει κανέναν εκτό. Σα ευχαριστώ. Ζήτω οι αγωνίστριε. Prego Παρακαλώ τους υποψηφίους προεδρούς να μιλούν λίγο πιο αργά, διότι οι διερμηνείς μεταφράζουν In questo Parlamento ognuno Εδώ στο Κοινοβούλιο ο καθής από εμά έχει δικαίωμα να εκφράζει τις ιδέες του, αλλά αν θέλετε να γίνεστε σεβαστοί θα πρέπει να σέβεστε και τους υπόλοιπους. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Νταβίτ Μαρία Σασόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Και εγώ είμαι υποψήφιος για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι υποψήφιος γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ισχυρή μόνο με ένα κοινοβούλιο το οποίο θα είναι σε θέση να διαδραματίσει ένα πιο σημαντικό ρόλο έχουμε να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικές προκλήσεις, οι οποίες ε, στο εγγύς μέλλον θα μας ε, δοκιμάσουν. Υπάρχει και η ίδια ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αμφισβητείται προκλήσεις τις οποίες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο αν παραμείνουμε ενωμένοι. Αν μπορέσουμε μέσω του σεβασμού της διαφορετικότητάς μας να ασκήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα νομοθετικά μας καθήκοντα, να ε, ελέγχουμε τον προϋπολογισμό, να κάνουμε έλεγχο και να δίνουμε πολιτικές κατευθύνσεις. Θέλω να είμαι ο εκπρόσωπος μαζί σας ε, των διαφορών μας και της ικανότητας λήψης αποφάσεων, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κεντρικό ρόλο, είναι αυτόνομο, έχει αξία η δημοκρατία την οποία εκπροσωπεί. Πρέπει λοιπόν όλοι όπως και να σκεφτόμαστε, να δεσμευτούμε προκειμένου να οικοδομήσουμε πραγματικά τον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ο οίκος της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Οι εκλογές ε, ήταν επιτυχής από πλευρά συμμετοχής. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς ε, που δεσμευτήκαμε ιδιαίτερα στις ευρωεκλογέ. διότι προσέφυγαν στις κάλπες για πρώτη φορά πολλοί ψηφοφόροι, πολλοί νέοι ψηφοφόροι και ακόμα και αυτή η συνέλευση ε, εκπροσωπεί αυτή την μεγάλη καινοτομία. Έχουμε 62% νέους ευρωβουλευτές, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό νέας ενέργειας. Οι ψηφοφόροι λοιπόν μας έχουν δώσει μια εντολή. Μας είπαν ότι πιστεύουν στο θεσμικό μας όργανο, ότι πιστεύουν στη δημοκρατία, στις ελεύθερες εκλογές και δεν μπορούμε εμείς να τους απογοητεύσουμε. Ε, από αυτό το κοινοβούλιο και από αυτή τη θητεία θα πρέπει λοιπόν να ε, καθοδηγήσουμε την ε, πιθανή και απαραίτητη αλλαγή ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και πιο σύγχρονη. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων. Και εδώ θα χρειαστεί όλη μας τη φιλοδοξία και όλο μας το σθένος, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της αλλαγής, της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής δικαιοσύνης της κυβέρνησης των μεταναστευτικών πολιτικών, την ε, ανάπτυξη, την εργασία και συνθήκων ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους. Εάν θέλετε να μου δώσετε την εμπιστοσύνη σας, ε, να προεδρεύσω, θα δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη για ένα κοινοβούλιο το οποίο θα είναι σύγχρονο, πιο διάφανο, ε, οικολογικά βιώσιμο και θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες θα ε, κάνω ό,τι μπορώ, θα αφιερώσουμε όλη την ευγένεια ώστε να γίνεται σεβαστό, να γίνεται σεβαστό το κοινοβούλιο από χώρε και από άλλα θεσμικά όργανα. Εσείς αγαπητοί συνάδελφοι βρίσκεστε εδώ διότι εκπροσωπείτε την ελπίδα. Ακόμα και την οργή των πολιτών μας, μην το ξεχνάμε κι αυτό, αλλά σίγουρα ε, τα συναισθήματα, την αίσθηση των ευρωπαϊκών λαών και εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, θα τίνω ευήκο στα όσα έχετε να πείτε, θα συνεργαστώ μαζί σας ε, με μεγάλη προσοχή, διότι αυτό σημαίνει ότι ανα πάσα στιγμή θα αφουγκράζομαι την αναπνοή και την ε, θέληση των γυναικών, των ανδρών και των νέων μας που έχουν εξαιρετικές ευκαιρίες ε, σε αυτή την Ευρώπη. Φανταστείτε ότι μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να ερωτευτούν χωρίς περιορισμούς θα είμαι θεματοφύλακας ε, της ανοιχτής αντιπαράθεσης, ε, της ε, πολυφωνίας και της άμεσης αντιπαράθεσης, αλλά πάντα σεβόμενη της απόψεις όλων. όλων εσάς και φυσικά και των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι εδώ, σε αυτή την Ολομέλεια, συχνά δεν το αντιλαμβανόμαστε, προστατεύουμε την ανεξαρτησία μας. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους Τίποτα δεν διαρκεί χωρίς τα θεσμικά όργανα. Πιστεύω ότι η έκκληση του Ζαμονέ ακόμα και σήμερα είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Ζάχρατηλ. Ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Για όσους ε, δεν με ξέρετε, είμαι ευρωβουλευτής από το 2004 και έχω δει πέντε πρόεδρους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη. Αυτό μου δίνει μια κάποια πείρα, ελπίζω, για να αντιληφθώ το τι θα μπορούσε να κάνει και τι πρέπει να κάνει αυτό το κοινοβούλιο, τι μπορεί να βελτιωθεί, τι μπορεί να αλλάξει και το τι πρέπει να κάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τι δεν πρέπει να κάνει. Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία επίσης μου λέει το ότι ε, καλό έναν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θεωρώ ότι ένας καλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι αμερόληπτος, ουδέτερος, μη κομματικός, θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες και όλους τους βουλευτές ισότιμα, ε, με δικαιοσύνη και με σεβασμό και ότι ο πρόεδρος θα πρέπει πάντα να θυμάται ότι δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του ή εαυτό της, αλλά το κοινοβούλιο στο σύνολό του. Και το τονίζω αυτό, στο σύνολό του είχα το πλέον πλεονέκτημα να ξεκινήσω την εκστρατεία μου λίγο νωρίτερα. Οπότε τύπωσα αυτό το φυλάδιο με τον ωραίο κύριο που βλέπετε. Ε, το έχετε ήδη λάβει μέσω email. Ελπίζω λοιπόν κάποιοι να είχατε την ευκαιρία να το διαβάσετε κιόλα. Μιλάω εκεί για το πώς θα ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα έχουμε ένα ανοιχτό και δίκαιο κοινοβούλιο, πώς θα ακούσουμε και θα ανταποκριθούμε στι ανησυχίε των πολιτών μα πώ θα έχουμε ένα κοινοβούλιο πιο αποτελεσματικό, με λιγότερη σπατάλη και πώ θα έχουμε μια στρατηγική εικόνα και όραμα για το μέλλον. Και πρώτα απ' όλα αναφέρομαι στις αρχές αυτές την αποκατάσταση της ισορροπίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ του ευρωπαϊκού επίπεδου και του εθνικού επίπεδου που μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και να βρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σταματήσουν οι εσωτερικές διαμάχες και να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας. Αναφέρω την ισορροπία και δεν θα πρέπει να ξεχάσω και μια άλλη πτυχή αυτής της ισορροπίας. Από το 2004, τα τελευταία 15 χρόνια, 13 νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 11 από αυτές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και εξ όσων γνωρίζω είμαι ο μόνος από αυτό το μέρος της Ευρώπης που είναι υποψήφιος για μία από τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζεται και αυτή η ισορροπία. Ένα τρίτο των κρατών μελών δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης και, εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος υποψήφιος για μία από τις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μία χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη και θεωρώ ότι χρειάζεται και αυτή η ισορροπία. Και τέλος, υπάρχουν μεγάλες χώρες αλλά και μεσαίες χώρες και μικρές και θεωρώ αν δεν κάνω λάθος, ότι πέρα από το Βέλγιο Είμαι ο μόνος εκπρόσωπος μιας μικρής ή μεσαίας χώρας που είναι υποψήφιος για μία από τις κορυφαίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ λοιπόν ότι χρειαζόμαστε και αυτήν την ισορροπία. Οπότε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με ψηφίσετε και σε αντάλλαγμα μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα αποτελέσω έναν καλό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ακούσαμε τους τέσσερις υποψηφίους για την Προεδρία, τις ιδέες τους ε, και τους λόγους για τους οποίους ζητούν την ψήφο σας. Πριν να περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας επιτρέπουν να μπορούμε να ελοποιούμε τις εργασίες μας με καλύτερο τρόπο, τους υπαλλήλους, τους βοηθούς, τους κλητήρες, τους διαρμηνείς. Γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως εκπρόσωποι του λαού και ευχαριστώ και τον Κλάους Βέλε, το Γενικό Γραμματέα και θέλω να το ευχηθώ χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενεθλιά του. Bene. Ora... Τώρα, να περάσουμε στην ελεύθερη επιλογή μας. Το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει θα εκλέξει τον πρόεδρό του ανεξάρτητα από εξωτερικές αιτιάσεις. Οι βουλευτές καλούνται να ψηφίσουν και να εκλέξουν τον πρόεδρό τους. Έτσι, όπως εξελέγην εγώ, με ελεύθερο τρόπο, είμαι πεπισμένος ότι και ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εκλεγεί με ελεύθερο τρόπο από όλους εσάς. Οι οδηγίες σε σχέση με την εκλογή του Προέδρου έχουν ε, σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές. Έχετε αντίτυπα στην είσοδο της αίθουσας. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1, για να εκλεγεί ένας υποψήφιος θα πρέπει να αποκτήσει στις πρώτες τρεις ψηφοφορίες την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων για να εκλεγεί θα πρέπει να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Τα λευκά ή τα άκυρα δεν ε, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των ψήφων. Τώρα, να περάσουμε στην ε, διανομή των ψηφοδελτίων και των φακέλων μέχρι την έναρξη της ε, ψηφοφορίας. Σας παρακαλώ να περιμένετε για να σας εξηγήσω το πώς ε, θα υλοποιηθούν οι εκλογές. Ε, έχουμε εκλέξει και τους ψηφολέκτες. Είναι όλοι εδώ, μου λένε ναι. Τώρα οι κλητήρες ε, μοιράζουν τους φακέλους ε, και τα ψηφοδέλτια. Για να ψηφίσει κανείς πρέπει να βάλει ένα σταυρό στο αντίστοιχο κουτάκι, στο κουτάκι που αντιστοιχεί στον υποψήφιο που επιλέγει. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο έναν ή μία υποψήφιο. Λοιπόν, αν θέλετε να διορθώσετε την ψήφα σας, μπορείτε να ζητήσετε ένα νέο ψηφοδέλτιο από το κλητήρα και θα δώσετε πίσω το λάθος ψηφοδέλτιο που θα καταστραφεί. Τώρα, αν ε, υπάρχουν ε, ε κάποια ε, λέξεις που έχετε γράψει ε, πάνω στο ψηφοδέλτιο, τότε ακυρώνεται. Επίσης, άκυρο θα θεωρηθεί αν ψηφίσετε πάνω από έναν υποψήφιο υπάρχουν και εκλογικές καμπίνες στην είσοδο του, της αίθουσας. στην κυκλίου, αν επιθυμείτε. Θα χρησιμοποιήσετε την κάλπη που ε, ουσιαστικά αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα του επιθέτου σας. Η πρώτη κάλπη είναι για τα α και β, η δεύτερη κάλπη από γ, δ, τρίτη κάλπη από ε έως g, τέταρτη από το H μέχρι το K, η επόμενη LM, η έκτη, E από το N ως το R, η έβδομη από το S ως το T και η όγδοη από το U ως το Z. Δεν μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι εγώ να ανακοινώσω ότι άρχεται η ψηφοφορία. Δεν θα καλέσω τώρα τους βουλευτές. Απλώς θα αναφέρω πότε αρχίζει και πότε κλείνει η ψηφοφορία. Τα ονόματα των βουλευτών που έχουν συμμετέχουν σε μυστική ψηφοφορία δημοσιεύονται στα πρακτικά και γι' αυτό το λόγο σας καλώ να υπογράψετε τον κατάλογο παρουσιών πριν να ε, βάλετε το ψηφοδέλτιό σας στην κάλπη. Να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να βάλετε το ψευδίλητο στην κάλπη που ανταποκρίνεται στο πρώτο γράμμα του επιθέτου σας. Πρέπει να δείξετε ή το badge ή την ταυτότητά σας στον ψηφολέκτη. Και καλό τώρα τους ψηφολέκτες ε, να μεταβούν στις αντίστοιχες κάλπες. La Άρχεται η ψηφοφορία.